είναι πάρα πολύ λυπηρά τα, όλες αυτές οι, οι ζωές που χάθηκαν και θα πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες αυτές και να τους μεταβιβάσουμε στις χώρες και στις οικογένειες στα συλληπιτήριά μας. 11 Μαρτίου αρχίζει στη Λιθουανία η 20η επέτειος της ανεξαρτησίας του. Πρόκειται για την επέτειο ανεξαρτησίας βεβαίως. Ήταν η πρώτη χώρα από το κομμουνιστικό μπλοκ που ε, κήρυξε αυτήν ανεξάρτητη. Έδωσε το σήμα, αν θέλετε, της κίνησης προς την ανεξαρτησία μεταξύ των μελών αυτής της περιοχής. 11 Μαρτίου ακόμη, το 1990, το Κογκρέσο της Εστονίας ενέκρινε ένα ψήφισμα σε σχέση με την ανεξαρτησία της χώρας αυτής μετά από 50 χρόνια κατοχής από τους Ρώσους. Συγχαίρω και τους Εσθονούς συναδέλφους, συνεπώς, για αυτή την επέτειο. 10 Μαρτίου τώρα έχουμε την επέτειο, την πεντηκοστή τη επανάσταση στο Θιβέτ, τη εξέγερση, μάλλον. Ζητούμε από τι κινέζικε αρχέ να μεταβάλουν τη θέση του προ του Θιβετιανού και να ξεκινήσουν διάλογο με τους Θιβετιανούς. Τώρα, μετά από τα σχόλια που έκανε ο κύριος Νάιτζελ Πάριτζ, ε, στην προηγούμενη Ολομέλεια σε σχέση με το 153.3 του κανονισμού επέβαλα μια κύρωση στον κύριο Φάρεντς Δέκα ημέρες diem είναι η κύρωση. Του αφαιρέθηκαν δηλαδή αυτά. Chciałem Państwa poinformować o innym wydarzeniu. Υπάρχει και ένα άλλο γεγονό για το οποίο θα ήθελα να σα ενημερώσω. Το εξή. Κλοπή. Κλοπή λοιπόν. Ένας από τους συναδέλφους της κλέψανε τα πράγματά της κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου των Βρυξελών. Έχοντας συζητήσει με τις βελγικές αρχές σχετικά. Η συνάδελφος κυρία Ντουρόν ενεργεί και σαν μεσολαβήτρια σε αυτές τις συνομιλίες που έχω και η κατάσταση έχει ως εξής. Μαζί με το Συμβούλιο, την Κομισιόν και εμείς θα θέλαμε να σχηματίσουμε μια ειδική ζώνη γύρω από τους ευρωπαϊκούς από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ζώνη ασφαλείας η οποία θα καλύπτεται από τις ομοσπονδιακές αρχές του Βελγίου. Έχουμε λοιπόν συνεχείς συνομιλίες, εντατικές μάλιστα, με τις βελγικές αρχές. Συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα και θα έχουμε επίσημη συνάντηση στις 20 Μαρτίου με την αστυνομία, με αυτό το στόχο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια γύρω από τα κτίρια του Ευρωκοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Ε, δεν αναφέρουμε μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο σε αυτή την περίπτωση. Προχωράμε. Περνάω στα πρακτικά της 25ης Φεβρουαρίου. Έχουν διανεμηθεί. Έχετε τυχόν ερωτήσεις σε σχέση με τα πρακτικά. Εάν όχι, εγκρίνονται.